πολύ. Η πρόεδρος, η κυρία Πακ, είναι στο Βερολίνο και δεν θα μπορέσει να παραστεί. Η πρώτη ε, αντιπρόεδρος η κυρία Τρίπελ είναι στο Ισραήλ άρα είμαι εγώ εδώ και σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση και άρχεται η συνεδρίαση καταρχήν αποδοχή της ημερησίας διατάξεως συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη σχετικά με το σημείο 6 Υπάρχει η πρόταση του κυρίου Μαρτίνες Μαρτίνες ο οποίος θα ε, έπρεπε να παρίσταται αλλά και αυτός έχει ένα πρόβλημα οπότε το σημείο αυτό δεν θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Εάν όμως δεν έχετε αντιρρήσεις ή διαφορετικές προτάσεις θα πρότεινα... Ε, και στα πλαίσια αυτά το 2011 έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος του Εθελοντισμού ούτως ώστε να υπάρξει συνειδητοποίηση του πόσο αυτές οι δράσεις αποτελούν και αυτές εκμάθηση πάρα πολύ χρήσιμη που βοηθά στις δεξιότητες, στις ικανότητες, στις δυνατότητες κοινωνίας και επίσης στηρίζει τις κοινέ ευρωπαϊκές ε, αξίες, την ελληνική δηλαδή και την κοινωνική συνοχή. Επίσης χρειάζεται περισσότερο να προσέξουμε το πώς θα ε, ε, αναπτύξουμε τις ικανότητες των διδασκόντων, αξιολόγηση, νέους τρόπους του πώς θα οργανώνεται αυτή η μάθηση. Επίσης εδώ τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ε, από να υπάρχει μια τέτοια ανάπτυξη των βασικών των δεξιοτήτων και όμως ε, δεν καλύπτονται όλες οι δυνατότητες από την επαγγελματική κατάρτιση γι' αυτό και θα πρέπει περισσότερο να προσέξουμε την γνώση των ξένων γλωσσών όσον αφορά τώρα το ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες δράσεις για τους μη προνομιούχους μαθητές μία μέθοδο που να είναι η πιο αποδοτική και φέτος άλλωστε είναι το έτος ε, κατά της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης και έτσι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να χτυπήσουμε τις ρίζες της ε, φτώχειας και μια τέτοια ε, εφαρμογή των μεθόδων της διαρκούς εκπαίδευσης να γίνει ολοένα και σε πιο μεγάλες περιόδους και αυτό να είναι κάτι που στο οποίο έχουν προσβασιμότητα όλες οι ηλικίε. Ανώτερη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Χρειάζονται νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας. Έτσι νομίζω ονομάζεται μία δράση και Επίσης χρειάζεται να βοηθήσουμε κάποιες ευκαιρίες για τους μαθητές για την ανώτερη εκπαίδευση. Επίσης χρειάζεται και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας να θεωρηθούν ότι πρέπει να προσεχθούν γιατί υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Θα πρέπει επομένω να βοηθήσουμε την κινητικότητα, οπότε σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να δούμε αυτές οι νέες δυνατότητες των διδασκόντων θα πρέπει να περιλάβουν τις νέες ανάγκες για τις νέες θέσεις εργασίας. Αυτό τονίζονται στην ε, έκθεση και ευχαριστώ όλους σας για τις παρατηρήσεις και σχόλιά σας εν κατακλείδε. Πρέπει να σας πω ότι εκρεμεί μία ε, διόρθωση η οποία αφορά την το, ισπανικό κείμενο, την ισπανική μετάφραση του κείμενου, το πρωτότυπο δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπαντία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση που κάνατε. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να ε, ξεκινήσουμε μια συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα συγκεκριμένες παρεμβάσεις αν ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Διάβασα με μεγάλη προσοχή την ε, πρόταση έκθεσης και νομίζω ότι πρόκειται για πολύ καλό κείμενο. Η έγκριση του κειμένου αυτού μάλιστα έρχεται σε μια ε, ιδιαίτερα δόκιμη στιγμή τη στιγμή δηλαδή που το Κοινοβούλιο ασχολείται με την στρατηγική 2020. Και είναι ευτυχής αυτή η σύμπτωση ή αυτός ο παραλληλισμός και καλό είναι να ληφθούν υπόψη, ε, να ληφθεί υπόψη και το κείμενο αυτό. Η πρόταση για την στρατηγική του 2020 υπογραμμίζει πολύ περισσότερο από ό,τι στη στρατηγική της Λισαβόνας την σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ακριβώς πρόκειται για έναν από τους πέντε κεντρικούς στόχους και πιστεύουμε ότι είναι ένας ιδιαίτερα ρεαλιστικός στόχος έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 10 χρόνια από τώρα να γίνει πιο ανταγωνιστική σε σχέση ε, με άλλες περιοχές του κόσμου, όπως ας πούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Επιτροπή στο δικό της έγγραφο, μεταξύ άλλων, προτείνει να φτάσουμε στο τουλάχιστον 40% των ε, φοιτητών που τελικά θα πάρουν το πτυχίο τους. Θα πρέπει επίσης να ε, κρατήσουμε κάτω από το 10% το ποσοστό ε, αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Και επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και την δυνατότητα μίας άτυπης ε, εκπαίδευσης, δηλαδή μίας εκπαίδευσης εκτός από το επίσημο σύστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως κάθε είδους εκπαίδευση να είναι ποιοτική. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί και αυτή η μη επίσημη εκπαίδευση που μπορεί να είναι και ευκαιριακή εκπαίδευση ακόμα. Ε, πιστεύουμε ότι μέσω της εκπαίδευσης θα μπορέσουμε να προωθήσουμε και τη διαδικασία της Κοπενχάγης που απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών. Στα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτύχαμε πολλά καλά ε, μέσω της μεθόδου της ανοιχτής συνεργασίας και του ανοιχτού συντονισμού και πιστεύω ότι πετύχαμε πολλά πράγματα. Επίσης, όσον αφορά τη διαδικασία της Μπολόνια, συμφωνώ με την Επιτροπή που λέει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο, αλλά όχι απλά να επενδύσουμε περισσότερο στα πανεπιστήμια, να επενδύσουμε καλύτερα και όχι να προσπαθήσουμε απλώς να βρούμε νέες πηγές ε, χρηματοδότησης ε, των, ε, ε της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των πανεπιστημίων δηλαδή, αλλά κυρίως να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε τα προγράμματα σπουδών, να τα ανακαινήσουμε κατά κάποιο τρόπο, να τα ανανεώσουμε, να τα προσαρμόσουμε στις νέες ανάγκες. Εάν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν θα λάμπουν τα πανεπιστήμια μας, δεν θα είναι τα καλύτερα στον κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει την ανταγωνιστικότητά της όσον αφορά τον τρίτο κύκλο σπουδών. Επίσης, στο ψήφισμά μας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ε, διάφορες ε, μορφές ε, κινητικότητας όπως το Εράσμους, το Marie Curie αλλά και το Grundig. Είναι ένας από τους τομείς που συχνά ξεχνάμε και το βλέπουμε μονάχα σαν κατάρτιση ενηλίκων και λίγο το αγνοούμε. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάρτιση των ενηλίκων συμπεριλαμβάνει τη διαβίου μάθηση. Υπάρχουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην, πολιτική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν ε, τα προσόντα έτσι ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας. Άρα θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Ε, άρα θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν περισσότερα προσόντα. Επομένως πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος. Έχουμε εδώ ένα ψήφισμα το οποίο έρχεται σε μια πάρα πολύ ε, σημαντική στιγμή. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι η ώρα που συζητάμε για τη στρατηγική 2020. Δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία. Τα επόμενα χρόνια, στην επόμενη δεκαετία, η εκπαίδευση θα παίξει πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι τα τελευταία δέκα. Άρα χρειάζεται και αισιοδοξία και αυτό, αυτή η αισιοδοξία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται εις την εργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ξεκίνησε καλά η συζήτηση, άρα ο κύριος Μπόρις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία επανέλαβε πολλές παρατηρήσεις τις οποίες είχαμε διατυπώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση και με τα μεγάλης χαράς διαπιστώνω ότι περιέλαβε αυτές τις παρατηρήσεις και τόνισε το πνεύμα το επιχειρησιακό, δηλαδή κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, μιλάει για τα πανεπιστήμια τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τον κόσμο της εργασίας. Μιλήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση πολύ και για τον αθλητισμό που είναι μια βασική δραστηριότητα για τους Ευρωπαίους σήμερα άρα και αυτό το στοιχείο περιλαμβάνεται στην έκθεση. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τον αθλητισμό είναι πολύ βασικές και το επαναλαμβάνω. Θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ότι όντως η έκθεση αυτή θα είναι πολύ σημαντική για την στρατηγική της Ευρώπης του 2020 διότι έπεται αυτής της στρατηγικής ε, και ε, θα καθορίσει την επιμόρφωση των Ευρωπαίων άρα ε, εδώ η παιδεία είναι ένα βασικό θέμα για να μπορέσει να προχωρήσει η Ευρώπη του 2020 και θα ήθελα να προτείνω κάτι ακόμη για να προσθεθεί στην έκθεση αυτή μιλάμε για τη συνεχή κατάρτιση, για, για την διαβίου μάθηση. Βεβαίως πάρα πολύ σωστά αναφερθήκατε στην διαβίου μάθηση δηλαδή προσχολική μετά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ήθελα όμως να τονίσουμε επίσης και τα άτομα που είναι πέραν των 45 ετών. Είναι μια σημαντική ομάδα όταν μιλάμε για διαβίου μάθηση, διότι τα άτομα μετά τα 45 σήμερα δεν βρίσκουν εύκολα εργασία, διότι η επιμόρφωσή τους έχει γίνει σε μια εποχή όπου οι σημερινές δεξιότητες δεν διδασκόντουσαν. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε αυτό το πέλεσιο ηλικία για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να ε, ξαναβρούν ε, εργασία ή τον ε, χώρο της εργασίας και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε και πάλι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία έχει κάνει εξαιρετική εργασία. Η κυρία Μπαντία Εκουτσέτ είναι μια πολύ ε, έμπειρη ε, ευρωβουλευτήνα οπότε δεν εκπλήσωμαι για την καλή της έκθεση. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ σε ένα σημείο Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να προσθέσει στην έκθεσή της για να συμπληρωθεί όσον αφορά τις διδακτικές, το διδακτικό προσωπικό διότι ε, ε, θεωρώ ότι πρέπει να τονίσει κανείς το διδακτικό προσωπικό αλλά ακόμη περισσότερο από ότι μέχρι τούδε διότι στην Ευρώπη έχουμε μία ενιαία αγορά. Εν τω μεταξύ έχουμε όντως μία ενιαία αγορά η οποία συναισθάθη και μπορούν οι εργαζόμενοι να διακινούνται ελεύθερα πέραν των συνόρων. Ξέρω όμως ότι στην Επιτροπή Πολιτισμού διαπιστώνουμε συνέχεια συνέχεια ότι ε, το ΑΕΠ πρέπει να αυξηθεί, ε, η αγοραστική δύναμη πρέπει να βελτιωθεί, ενώ υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Για να μπορέσουμε λοιπόν όντως να βελτιώσουμε το επίπεδο ευημερία θα πρέπει να προετοιμαστούμε ε, σε καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση και αυτό εξαρτάται από την βασική εκπαίδευση και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε καλή βασική εκπαίδευση με το να έχουμε ε, επαρκές ε, καλό διδακτικό προσωπικό. Πώς θα το επιτύχουμε με καλή εκπαίδευση και κατάρτιση του ε, εκπαιδευτικού προσωπικού. Για να υπάρξει λοιπόν αυτή η εκπαίδευση πρέπει να τους θεωρήσουμε σαν ένα σημείο πυρήνα για την προσπάθεια που καταβάλουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί ακόμη περισσότερο και για να γίνει αυτό χρειάζεται μια στρατηγική από την πλευρά της ε, Επιτροπής για την κατάρτιση του προσωπικού διότι πολλές φορές μιλάμε πολύ για αυτό το θέμα αλλά πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή όντως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να περάσουμε από, τις, ε, από τα λόγια στις πράξεις και στην Ευρώπη θα πρέπει να ε, προχωρήσει η καλύτερη κατάρτιση του εκπαιδευτικού δυναμικού και αυτό είναι ένα σημείο που θα ήθελα να τονιστεί περισσότερο στην έκθεση της κυρίας Μπαντία. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τάκουλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και στην εκπαίδευση. Ξέρει πολύ καλά περί τίνο πρόκειται και ξέρει γιατί μιλάει. Είναι δάσκαλο. Σε μια τάξη βεβαίως έχουμε, ε, δασκα... έχουμε τους μαθητές αλλά έχουμε και δάσκαλο. Και ο δάσκαλος είναι εκεί και για λόγους ε, εφαρμογής της πειθαρχία, αλλά και για να κινητοποιήσει τους μαθητές του, ε, για να κάνει ελκυστική τη διδασκαλία του και το αντικείμενο της διδασκαλίας του για τα παιδιά, για τους μαθητές του. Ξέρουμε ότι έχουμε πολύ διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και πολύ διαφορετικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό ε, θέλουμε σιγά σιγά να απαλληθεί. Πολύ ωραία λοιπόν, όλα αυτά περιέχονται στην έκθεση της κυρίας Μπαντία Ο επόμενος είναι ο κύριος Σμιτ, παρακαλώ. Και μετά Σάντσε Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω στα Ουγγρικά. Ναι, ναι, συνεχίζω στα Ουγγρικά. Ε, σας ευχαριστώ, έλεγα και επίσης συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Είναι πάρα πολύ σωστό το ότι κάθε τόσο αναθεωρούμε και ξανασυζητούμε τι γίνεται με την ισόβια εκμάθηση από το ε, νηπιαγωγείο μέχρι την αποφύση από το πανεπιστήμιο και στη συνέχεια. Θα ήθελα κάτι να πω, με έχει καλύψει ένα σημείο ο συνάδελφος Μπόρε, διότι ανέφερε ότι η προετοιμασία, η, η ηλική, η πιο σωστά η φυσική αγωγή πουθενά δεν εμφανίζεται. Δεν θέλω να πω ότι δεν αρέσει ο αθλητισμός στην κυρία Μπαδία. Όχι θέλω να πω ότι το 60% των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουν κανένα σπορ, κανένα. Οπότε έτσι είναι πιο εύκολο να αρρωστήσουν. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει στο μέλλον. Θα πρέπει αυτό να γίνει μάθημα, μάθημα βασικό. Θα πρέπει επομένως να προετοιμάζεται το παιδί για το τι θα γίνει όταν ε, ενηλικιωθεί και επομένως ε, να ετοιμαστεί για την ώρα του αθλητισμού. Οπότε, ακόμα και στους παιδικούς σταθμούς θα πρέπει να υπάρχει κίνηση, φυσική αγωγή. Ε, στο γυμνάσιο. Θα πρέπει να υπάρχει σαν υποχρεωτικό μάθημα η γυμναστική. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ βασικό μάθημα. Είναι κάτι το απαραίτητο. Μια που μιλάμε για τον αθλητισμό, θα σας πω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε κατά πόσο γίνεται ε, να αξιολογήσουμε με αριθμούς τα, τα, τα, τα μαθήματα, τις ε, δεξιότητες, τα προσόντα δηλαδή, να δούμε για τα 8 βασικά μαθήματα τι βαθμοί έχουν δοθεί. Αυτό όμω θα γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν λοιπόν κάποιο τελειώνει τι σπουδέ του, τότε να μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση. Φυσικά και θα είναι εφικτό να βρούμε μια μέθοδο αποτίμηση και αξιολόγηση. Επομένω, σα επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει μεταξύ των βασικών μαθημάτων να βάλουμε και τη γυμναστική. Αν θέλουμε να μπορούν να είναι και σωματικά και πνευματικά ικανά και δυνατά τα παιδιά μα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την κυρία Μπαδία για την έκθεσή της σε συνέχεια των όσων μας είπε ο κύριος Σμιτ και εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι που μου φαίνεται ότι δεν αναφέρθηκε, δεν εξαντλήθηκε. Ε, στην ε, εισήγηση της κυρίας Μπαδία είναι όσον αφορά τα πολιτιστικά γιατί είπαμε για τον αθλητισμό, είπαμε για την φυσική αγωγή, όμως από την άλλη μεριά τα καλλιτεχνικά, τα πολιτιστικά θα πρέπει και αυτά από μια μικρή ηλικία να είναι τμήμα της ε, παιδείας ούτως ώστε να μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητες του το παιδί και πέρα από το όριο του σχολείου και να είναι δυνατόν καθόλου τον τρόπο από την προσχολική ηλικία ή από τον παιδικό σταθμό μέχρι το, μέχρι το τέλος της ε, εκπαίδευσης και άλλωστε ε, αυτά, ε, αυτά τα καλλιτεχνικά βοηθούν και στα άλλα μαθήματα είναι η κληρονομιά, η πολιτιστική, το περιβάλλον γιατί νομίζω ότι οι δυσκολίες στο σχολείο μπορούν να ξεπεραστούν και επομένως θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το σημείο, μια που δεν έχει ενταχθεί ε, η τέχνη, τα πολιτιστικά στα βασικά μαθήματα, ενώ νομίζω ότι είναι σημαντικό και χρειάζεται από κάθε πλευρά στη εκπαίδευση και στην παιδεία. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν φαίνεται να ζητάει κάποιος άλλος βουλευτής το λόγο και επομένως τρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει πρόσωπος της Επιτροπής ε, που θα ήθελε να πάρει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την στήριξη η οποία εκφράζεται στην έκθεση, την ε, έκθεση που έχει προετοιμάσει η κυρία Μπαντία και αντιλαμβάνομαι και ερμηνεύω ότι αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σας ε, ικανοποίησε και θέλετε να τονίσετε διάφορα θέματα. Βεβαίως είναι πολύ βασική η έκθεση αυτή για τις, ε, ε, για τις αρμοδιότητες κλειδιά ε, και ιδίως όσον αφορά τη διαβίου μάθηση και τη συνεχή μάθηση είναι βασικό να προετοιμάζει κανείς τους ανθρώπους από την προσχολική εκπαίδευση κατά την σχολική εκπαίδευση στην επαγγελματική κατάρτιση όχι μόνο για τα επαγγέλματα όπου θα πρέπει κανείς να καταρτήσει αλλά στα θέματα που ανέφερε ο κύριος Σμιτ. Δηλαδή η πολιτιστική επιμόρφωση είναι επίσης ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναπτύσσεται για να μπορέσουν οι άνθρωποι να προσαρμοστούν στην αγορά εργασίας και να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία ε, και για τα πανεπιστήμια. Όπως το είπε και η κυρία Μπαντία είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχουν αυτές οι εγκάρσιες αρμοδιότητες αρμοδιότητες, η περαιτέρω κατάρτιση ε, που είναι πολύ χρήσιμες. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας και τονίζω αυτά τα οποία ελέγχθησαν σχετικά με την ε, ε, σχέση εις τον χώρο της εργασίας με την ευρύτερη στρατηγική για το 2020. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, στρέφουμε τώρα προς την κυρία Μπαντία. Θέλετε να πάρετε το λόγο έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για την ε, έκθεσή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όλους για τις παρατηρήσεις που υποβάλλατε. Και εγώ κράτησα κάποιες σημειώσεις όσον αφορά τη στρατηγία το 2020. Μου φαίνονται πάρα πολύ εύστοχα το ότι θα πρέπει να αναφερθεί η σχέση μου που έχει αυτή η έκθεση με τη στρατηγική του 2020. Νομίζω πως είναι ενδιαφέρον σε κάποια ιδεολογική έκθεση κάπου σε μια παράγραφο να τονίσουμε τη σχέση αυτών που λέμε τώρα με την ε, θα δει το 2020. Όσον αφορά τώρα για το επιχειρηματικό πνεύμα, τη σχέση με τον κόσμο της δουλειάς, τον επαγγελματικό βίο, ε, την τελευταία φορά, τέλος την πρώτη φορά που κάναμε την ε, ανταλλαγή απόψεων, το άκουσα που το είχατε πει και θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα αυτά, όπως και αυτό που είπε ο κ. Σμιθ για τον αθλητισμό. Άμα ξεχάσω να γράψω κάτι να μου το θυμίσετε, γιατί επί της ουσίας συμφωνώ ότι θα πρέπει ο αθλητισμός να καλύπτεται από την ε, παιδεία. Κύριε Τακούλα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και έχει σημασία το ότι προέρχεστε από τη Φιλανδία, που είναι χώρα που πάντοτε αναφέρουμε ως μια χώρα που έχει τις καλύτερες επιδόσεις στην παιδεία, στην κατάρτιση. και με την ευκαιρία θα πρέπει και στον κύριο Σάντζας να απαντήσω ότι η κατάρτιση των καθηγητών, των διδασκόντων, όλα, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ίδια τα έχω αναλάβει. Γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και συμφωνώ και μαζί σας ότι πρόκειται για πολύ βασικά ζητήματα και μαθήματα, αλλά και όσον αφορά τα πολιτικά και τα καλλιτεχνικά που θα πρέπει να εισαχθούν από τη, τη, τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Αυτό θα πρέπει να γίνει γιατί έτσι ε, αξιοποιείται η, η πολιτική παράδοση, αξιοποιείται η, η δημιουργικότητα που έχουν τα παιδιά από πολύ μικρά. Γι' αυτό και συμφωνώ μαζί σας σε όσα είπατε. και για την εκπαίδευση των ε, διδασκόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προσθέτω ότι η βελτίωση αυτής της εκπαίδευσής τους έρχεται και δένει με το κοινωνικό τους κύρος με το οποίο θα πρέπει να τους θωρακίσουμε αν θέλουμε να δουλεύουν σωστά στις τάξεις των σχολείων. Και βέβαια και σύμφωνα με αυτό το οποίο είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενο της ανακοίνωσής της. Νομίζω ότι σιωπηρά όλοι συμφωνούμε ότι η κατάρτιση, η παιδεία είναι το κλειδί του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό και συμφωνούμε όλοι. Όμως θέλω να ζητήσω κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με απασχολεί αυτό. Το πώς θα βελτιώσουμε την ε, κατάρτιση των διδασκόντων γιατί στο στρατηγείο του 2020 λέμε για, τους, για τις καινούργιες προκλήσεις, την καινούργια οικονομία, την κρίση, την πράσινη οικονομία, τη λευκή οικονομία. Νομίζω θα πρέπει να δούμε τι χρειαζόμαστε. Τι κατάρτιση χρειάζεται για την νέα οικονομία ο κόσμος. Και έτσι αντίστοιχα και εμείς να δούμε πώς θα εκπαιδεύσουμε τους καθηγητές, τους διδάσκοντες. Ευχαριστούμε πολύ και στρέφουμε ακόμα μια φορά προς τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν αν θέλει να απαντήσει, αν θέλει να σχολιάσει τα λεγόμενα της κυρίας Μπαντία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την ερώτηση. Το σημείο κινήσεως εδώ έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες ε, ε, κλειδιά εγκαρσίως δηλαδή στον τομέα της ε, επιμόρφωσης ε, και ε, περαιτέρω κατάρτισης των διδασκάλων για να μπορέσουν να βελτιωθούν οι δεξιότητες που είχαν παραμεληθεί μέχρι στιγμής Είχαμε κάνει μία ειδική ε, κοινοποίηση ανακοίνωση όπου λέγαμε ότι οι ε, ε, δεξιότητες που αναφέρονται στο διδακτικό πρόγραμμα υπάρχουν μόνο στο χαρτί και θα πρέπει να μεταδίδονται από τους διδασκάλους ή στους εκπαιδευόμενους. Αυτή είναι λοιπόν μία από τις δεξιότητες τις οποίες θέλουμε να προωθήσουμε στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και θα ήθελα κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε προς ε, τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ε, δεν ξέρω αν ε, μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, γι' αυτό και συμφωνώ ότι το θέμα αυτό της καταρτήσεως των διδασκάλων είναι σημαντικό και θα πρέπει να συναντηθούμε με τα κράτη-μέλη και να προωθήσουμε την προτεραιότητα αυτή που είναι η επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, για τις αποσαφηνήσεις σας και γενικότερα για την συζήτηση. Επί της εκτέσεως αυτής υπάρχει προθεσμία υποβολής τροπολογιών ε, και είναι η 26η Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Πρόκειται για μια ημέρα Παρασκευή. <clears throat> Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το θέμα της κυρίας Μπαντία. Φτάνουμε επομένως στο επόμενο σημείο, είναι το σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως. και προβλέπει η ανταλλαγή απόψεων για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ε, για πέστε μας κυρία Μπραντς, περί πρόκειται ακριβώς. Πρόκειται για ένα θέμα ε, πληροφοριακό απλώς ε, ή θα γίνει συζήτηση. Α, μάλλον όχι. Έτσι κι αλλιώς μετά στη διάρκεια της συνεδρίας των συντονιστών θα δούμε ποιος θα ασχοληθεί με την ε, έκθεση αυτή. Επομένως τώρα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Επί της διαδικασίας αποσαφηνίζω ότι θα δώσουμε πρώτα απ' όλα το λόγο στους καλεσμένους μας. Μετά θα θέσουμε ερωτήματα και θα κάνουμε σχόλια Κυρία Μπραντς, παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Η πρόταση αυτή της 9ης Μαρτίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εισάγει στην Ευρώπη το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πρόκειται για απόφαση Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βασίζεται στο άρθρο 167 της Συνθήκης. Πρόκειται για άμεση απάντηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του 2008 που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με πρόταση σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, θα ήθελα να κάνω μια γενική εισαγωγή στην πρόταση και να πω σε γενικές γραμμές πώς εμείς ε, προτιθέμεθα να επιλέξουμε τις τοποθεσίες γιατί διαφοροποιείται αυτή η πρωτοβουλία από άλλες υφιστάμενες ε, πρωτοβουλίες και κάποια άλλα σημεία κλειδιά. Πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο στόχος, ο σκοπός αυτής της πρότασης η ιδέα είναι να δοθεί το σήμα σε περιοχές οι οποίες ε, παρουσιάζουν σημαντική συμβολική αξία ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι θεμελία λήθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, για να μάθουν οι πολίτες, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, που βασίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βεβαίως ε, ευελπιστούμε και σε αύξηση του, της προσέλευσης τουριστών και της επισκεψιμότητας των τοποθεσιών αυτών. Επομένως, θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις. πώς θα γίνεται η επιλογή. Ανοιχτές θα είναι τοποθεσίες από τις 27 χώρες μέλη σε εθελούσια βάση. Κάθε χώρα μέλος θα, έχει ε, ίσες ε, δυνατότητες και ευκαιρίες να ε, προτείνει έως δύο τοποθεσίες για τις οποίες θέλει το Σύμμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα υπάρξει δηλαδή μια εθνική προεπιλογή. Μετά μία ομάδα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων ε, θα προτείνει μία ε, τοποθεσία σε κάθε χώρα μέλος που τελικά θα λάβει το σήμα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ε, τελικά το πολύ 27 τοποθεσίες που θα πάρουν το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινωνίας κάθε χρόνο σε σχέση τώρα με υφιστάμενες άλλες ε, πρωτοβουλίε, θα ήθελα να επιστήρω την προσοχή σας ότι ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ε, πρόταση αυτή έτσι ώστε να μην υπάρξουν επικαλύψεις ε, με άλλες διαδικασίες οι οποίες υφίστανται ήδη είτε από την UNESCO είτε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό είναι απολύτω θεμελιώδε και για εμά και για τι χώρε μέλη βέβαια, να αποφευχθούν οι επικαλύψει. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του σήματος που το ξεχωρίζουν από άλλες πρωτοβουλίες. Πρώτα απ' όλα, το σήμα αυτό θα δίδεται σε τοποθεσίες οι οποίες έχουν παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουν δηλαδή ε, ένα ιδιαίτερο ευρωπαϊκό θυμικό, να παίξουν ρόλο στο, ιδιαίτερο ευρωπαϊκό θυμικό. Δεύτερον, δεν αναφερόμαστε μονάχα στην ομορφιά ή μάλλον δεν αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην ομορφιά ή στην αρχιτεκτονική αλλά στη σημειωτική ε, και στους συμβολισμούς ε, της τοποθεσίας. Ε, τρίτον, μας απασχολεί περισσότερο η εκπαιδευτική δυνατότητα που δίνεται κυρίως στους νέους. Τέλος, αυτό το σήμα θα γίνει πιο αποτελεσματικό μέσω δικτύωσης. από πού προέρχεται η πρόταση αυτή και γιατί τα κράτη-μέλη ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με την ε, πρόταση αυτή. Η αρχική ε, σύλληψη ε, ξεκίνησε το 2005 μετά από μία σειρά αρνητικών προσήμων λόγω των αρνητικών εκβάσεων των δημοψηφισμάτων εκείνη την εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργήσε μια κακή εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως το σήμα αυτό ε, στόχο είχε να μικρύνει την απόσταση που είχε και τα χάσματα που είχαν δημιουργηθεί τον Απρίλιο του 2006 σε καθαρά διακυβερνητική βάση και χωρίς ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε μια πρώτη προσπάθεια ε, για το σήμα αυτό και σήμερα 17 με κράτη-μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και έχει δοθεί το σήμα σε 64 περιοχές ή τοποθεσίες. Όμως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συγγνώμη, τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν σε αυτήν, συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία ε, είδαν ότι υπήρχαν ελλείψεις και δυσκολίες και γι' αυτό προσέτρεξαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να απαλληφθούν οι δυσκολίες και οι ελλείψεις αυτές. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε σαν καθαρά διακυβερνητική και ε, προχώρησε για να αποκτήσει το ευρωπαϊκό πρόσημο. Τώρα, πώς ε, προετοιμάστηκε η διαδικασία αυτή. Μετά από τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο το 2008, ε, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση συμπεριλαμβανομένων ε, δημοσίων συναντήσεων, αλλά και online ερωτηματολογίων. Ξεκίνησαν επίσης μελέτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων όλα αυτά κατέδειξαν ότι το σήμα έχει ισχυρό δυναμικό και ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια διαδικασία με πραγματικά προστιθέμενη αξία και μπορεί να έχει έναν ουσιώδη αντίκτυπο. Θα ήθελα τώρα να σας να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία κλειδιά. Τα κριτήρια είναι σαφή, απλά βασίζονται ε, ακριβώς στην ε, ε, ευρωπαϊκή σημασία της τοποθεσίας, στις δραστηριότητες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές οι οποίες προσφέρονται και την ορθή διαχείριση της τοποθεσίας είναι τέτοια ε, η διαδικασία ε, προεπιλογής και επιλογής που μονάχα οι τοποθεσίες οι οποίες πραγματικά συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν και να λάβουν το σήμα. Βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρξει και έλεγχος και εποπτεία ε, καθ' όλη την διάρκεια της ε, διαδικασίας έτσι ώστε ακόμα και μετά να συνεχιστεί η εποπτεία αυτή και οι τοποθεσίες οι οποίες έχουν πάρει το σήμα να εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο ύψος του σήματος αυτού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει διαδικασία κύρωσης και επομένως αφαίρεσης του σήματος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Κάθε έξι χρόνια εισάγεται ε, η έννοια της εξωτερικής, του εξωτερικού ελέγχου ε, από ανεξάρτητη αρχή. Όσον αφορά τώρα τον προϋπολογισμό, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πολύ, μικρή, μικρός θα είναι ο αντίκτυπος στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το μόνο κόστος το οποίο θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορά το κόστος του Ευρωπαϊκού Συντονισμού, της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής ε, ε, διαδικασία, τη λειτουργία του πάνελ των εμπειρογνωμόνων, το networking και κάποιες, κάποιους ανθρώπινους πόρους που θα απαιτηθούν από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως μέσα από την αναμόχλευση των κονδυλίων θα βρεθούν ε, οι απαραίτητοι πόροι. Κατά τα λοιπά πρόκειται για εθνικό θέμα και θα καλύπτεται από εθνικού προπολογισμού. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να υπάρξει μια αρχική διετής μεταβατική περίοδος μετά τη θέση σε ισχύ της απόφασης. Ε, η ιδέα είναι δηλαδή ότι ε, τον πρώτο χρόνο οι τοποθεσίες ε, θα μπορέσουν να προσαρμοστούν ε, από το παλιό καθεστώς στα νέα κριτήρια έτσι ώστε να ε, λάβουν το νέο σήμα και Επίσης, τα κράτη-μέλη τα οποία δεν συμμετέσχουν στην προηγούμενη πρωτοβουλία να έχουν την δυνατότητα να προτείνουν μια πρώτη σειρά τοποθεσιών πριν ξεκινήσει η πραγματική κανονική διαδικασία προεπιλογής και επιλογής, έτσι, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Εν συμπεράσματι, ε, βασιστήκαμε σε διάφορες αρχές προετοιμάζοντας την πρόταση. Πρώτον ε, είναι ε, να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται περισσότερα από τα αιτήματα των περισσότερων κρατών μελών και να είναι όσο γίνεται πιο συνενετική η πρόταση αυτή. Δεύτερον, θελήσαμε να δώσουμε, να αναλάβουμε πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες καινούργιες οι οποίες θα παρουσιάζουν βελτίωση και σαφή, ε, σαφώς καλύτερη προστιθέμενη αξία από προηγούμενες προτάσεις. Ε, σεβαστήκαμε την αρχή της επικουρικότητας. Ε, τέταρτον, θελήσαμε ένα σχήμα το οποίο ε, θα είναι όσο γίνεται πιο απλό στη διαχείρισή του αλλά και όσο γίνεται πιο ελκυστικό ε, στην ε, πραγμάτωσή του. Τέλος, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε μία ε, εξαιρετικά ορατή πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε ότι το καταφέρουμε. Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω οποιασδήποτε ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την εισήγησή σας, κυρία. Και τώρα, επανερχόμαστε στην συζήτηση. Άλλωστε, βλέπω ότι τα είπε όλα η Κομισιόν, κανείς δεν έχει να προσθέσει. Α, έχει το λόγο κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σύγκρισή τη, γιατί τώρα Έχουμε κάτι το πάρα πολύ συναρπαστικό μπροστά μας, δηλαδή θα πρέπει να κάτσουμε και να ε, αξιολογήσουμε το πώς έχει η κατάσταση της πολιτικής οικονομίας στην Ευρώπη, γιατί δεν μιλούμε για ένα συγκεκριμένο μέρος, ε, για ένα συγκεκριμένο σημείο, πρόκειται για μια προσωπικότητα, πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα, ένα έργο, όμως έχουμε, έχουμε τελικά και κάποιες πόλεις, έχουμε κάποιες ε, καθορισμένες ε, περιοχές, μικρές περιφέρειες ε, και αυτό με χαροποιεί γιατί βλέπω ότι όλα αυτά αποκτούν κάποια προσωπικότητα ε, έχουν τη σφραγίδα την ευρωπαϊκή δεν θέλω να, να, να, να προσβάλλω κανένα ούτε με Πολωνός όμως νομίζω ότι θα έπρεπε να δοθεί ένα βραβείο στον Σοπέν Ούγκρος είμαι, δεν είμαι Πολωνός, παραλαμβάνω. Και επομένω θα πρέπει αυτό να γίνει όταν να προβληθεί η ευρωπαϊκή κοινωνιά. Μετά λέμε για μια πόλη. Εντάξει, καλό και αυτό, πάρα πολύ συναρπαστικό και τελικά ο στόχο είναι να ελκύσουμε τον τουρισμό και έτσι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πανευρωπαϊκό, ούτω ώστε αν μια μέρα έρθει ένα Ιαπωνέζο, ένα Ινδό εδώ στην Ευρώπη, κάποιο από κάπου μακριά, να μπορεί να κάνει αυτή τη διαδρομή στι πόλει δηλαδή, τον, τον, τον, που συναποτελούν αυτό το, το, το δίκτυο. Κοιτάξτε τώρα να δούμε πώς θα, ε, πώς θα αυτή η επιτροπή που θα αποφασίσει. Και πώς θα, τι, τι κυκλική αλλαγή θα γίνει, αυτή η σφραγίδα, αυτό το σήμα, θα κρατάει για ένα χρόνο. Μα τότε, τότε θα έχουμε για όλη μας την κληρονομιά ένα μέλλον Όχι, θα πρέπει ένα, ένα, ένα σήμα Α, ένα, ένα, ένα ένα, ένα λέτε. Α, ωραία. Α, αυτό εννοούσατε. Εντάξει. Ωραία. Το, α, τότε είναι ακόμα πιο μεγάλη πρόκληση. Αλλά να δούμε πώς θα συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή, τι, τι, μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι και το ποσοτικό στοιχείο. Εδώ δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις α, χρησιμοποιώ έναν οδηγό Michelin για να δώσει ποιο εστιατόριο θα πάω να φάω. Και ποτέ δεν κάνει λάθος ο οδηγός Michelin. Έχει τόσο αυστηρά κριτήρια ούτω ώστε ε, για να πάρει κανείς ένα και μόνο αστέρι θα πρέπει χρόνια χρόνια να, να, να δουλεύει με συνέπεια και γι' αυτό και ο κόσμος εμπιστεύεται τους οδηγούς Michelin. Και όσο πιο καλό είσαι, πιο πολλά αστέρια Michelin παίρνεις. Άρα τι θα έχουμε, ε, σε αυτή την Επιτροπή έναν από κάθε χώρα μέλος. Θα υπάρχουν ίσως ε, κάποιος αντιπροσωπεύει κάποιον άλλο. Τι θα γίνει. Ο Πρόεδρος. Έχει το λόγο. Κυρία Χάνι Μπολ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρόταση αυτή, η οποία μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά τα πράγματα αυτά δεν είναι εύκολα στην αρχή και παρόλο που υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να προτείνουμε μη μεταβατική περίοδο, διότι ελπίζουμε ότι αυτό σημαίνει ότι ε, θα μπορέσουν ε, να εμπλακούν και τα κράτη τα οποία υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο, δεν ξέρω καν ποια είναι, αλλά θα μπορούσαν να ε, πιστούν να ενεργήσουν. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ε, χρηματοδότηση προέρχεται από τα κράτη-μέλη και απλούστατα θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά ε, θα ε, διατεθούν διότι ε, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οποία ακούσαμε ε, θα είναι μια κυβερνητική ε, πρωτοβουλία κάτι που είναι τελείως διαφορετικό από, την, από, τα πολιτιστικά θέματα που προέρχεται από τα κράτη που αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό το θέμα αυτό είναι για αυτά. Εδώ μιλάμε για ιστορικά μέρη τα οποία χρειάζονται διαφορετική εμπλοκή. Εάν έχω δίκιο, σας παρακαλώ να μου το επισημάνετε. Θα ήθελα να ακούσω ποιες είναι οι εναλλακτικές προτάσεις επ' αυτού. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν πολλά για να εξασφαλίσουν ότι ε, έχουν πληρωθεί τα δέοντα και υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση χωρίς να υπάρχει ε, συγκέντρωση σε ορισμένα κράτη-μέλη και ουσιαστικά το, κίνητρο το να περιληφθεί και ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο προχωρά. Ε, γι' αυτό και νομίζω από πλευράς πολιτιστικής είναι πάρα πολύ καλό και θα συμφωνούσα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και ορισμένες ε, πρακτικές λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να διευκρινιστούν. Ευχαριστώ κυρία Χάνιμπαλ. Οπότε τώρα έχω την κυρία Σάντσε Σμιτ, μετά τον κύριο Παπα-Νικολάου, αλλά καταρχήν η κυρία Σάντσε Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επέμβω σε διάφορα σημεία. Νομίζω ότι είναι βασικό να καθορίσουμε συγκεκριμένα για όλα τα κράτη-μέλη τι εννοούμε όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή κληρονομιά, για να μην υπάρξει σύγχυση με άλλες επικεφαλίδες. Μετά θα ήθελα να ξέρω αν έχουμε αλλάξει ε, γνώμη όσον αφορά τις ε, συγκεκριμένες ε, προτάσεις ε, για να υπάρχει ευρωπαϊκή εμπλοκή και θα έπρεπε όλες οι ιστοσελίδες, όλα τα σημεία τα οποία θα λάβουν αυτή την σήμανση ε, συνεπιφέρεται μια συγκεκριμένη σημασία. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε σημασία στο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει ε, το κάθε κράτος σε έναν χώρο, σε μία ιστοσελίδα. Δηλαδή ε, θα πρέπει να υπάρχει και παιδαγωγική και ε, εκπαιδευτική και να μην είναι μόνο τουριστική, τουριστικό διάβημα αλλά να είναι επιμορφωτικό. Ευχαριστώ. Ο Στογιάννοφ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Όντως η ιδέα του, της Επιτροπής είναι εξαιρετική. Έχω πολύ θετική αντιμετώπιση και θα ήθελα να περιλάβουμε και ένα πιο πρακτικό στοιχείο. Παραδείγματο χάρη, εάν αύριο γυρίσω στην εκλογική μου περιφέρεια και τους πω περί αυτών επειδή η εκλογική μου περιφέρεια είναι η πόλη του Πλόφτιφ η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Βουλγαρία αν τους μιλήσω για αυτή την πρωτοβουλία φοβάμαι ότι τα άτομα τα οποία θα καταρτήσουν τις υποψηφιότητες θα θεωρήσουν ότι είναι κάτι πολύ αφηρημένο και θα μας ρωτήσουν τι μέλη εάν εμείς κερδίσουμε ε, και επιτύχουμε να πάρουμε αυτό το σήμα. Θα πρότεινα λοιπόν το εξής. Πέραν ε, να συμπεριληφθεί στις 27, ε, στις 27 επιλογές να υπάρξουν και, και άλλα κίνητρα πρακτικά, ρεαλιστικά υλικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι θα κερδίσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ σημαντική και εγώ προέρχομαι από μια χώρα που έχει μεγάλη ιστορία και ε, πολιτιστικά μνημεία παγκοσμίου αναγνωρισιμότητας. Ε, το ερώτημα είναι παραπλήσιο και από την πλευρά μου με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Ε, συζητάμε εδώ και ε, αποφασίζουμε για τα κριτήρια και τον τρόπο με τον οποίο θα αποδίδουμε αυτό το σήμα ε, στα, ε, στα διάφορα πολιτισμικά μνημεία. Και η ερώτηση και δική μου προς την Επιτροπή είναι αυτή. Αφού έχουμε αυτή την, αυτή τη σήμανση σε όλα τα κράτη-μέλη και σε διάφορα πολύ σημαντικά μνημεία στα πλαίσια του συντονισμού, στα πλαίσια της επικουρικότητας καταρχάς από πλευράς ε, επιτροπής που, και της επικουρικότητας και την εθελοντική βάση πάνω στην οποία θα κινηθούν τα κράτη-μέλη και στα πλαίσια του συντονισμού που θα υπάρχει από την πλευρά της Ευρώπης υπάρχουν πιο συγκεκριμένες προτάσεις και ενδεχομένως δράσεις και στο επίπεδο της προβολής και στο επίπεδο ε, του διαλόγου, του διαπολιτισμικού μεταξύ των κρατών μελών πιο συγκεκριμένα προκειμένου αυτή η σήμανση συνέχεια να έχει και απτά αποτελέσματα τα οποία και εμείς θα μπορούμε να παρουσιάζουμε στους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, τώρα έχουμε μία σειρά από ερωτήματα που έχουν τεθεί και σχόλια τα οποία έχουν γίνει. και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ναι, θα απαντήσω σε διάφορες ε, ερωτήσεις, όπως ας πούμε αυτό που ε, η πρώτη που ετέθη σχετικά με προσωπικότητες ή τον Σοπέν. Ναι, ε, το σήμα προβλέπεται βάσει του άρθρου 2 της πρότασης για, αναφέρεται μάλλον σε απτά συγκεκριμένα ε, σημεία, ε, γεωγραφικές περιοχές συγκεκριμένες. Όμως ε, η οποιαδήποτε μη απτή άειλη πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ληφθεί υπόψη βάσει αυτής της πρωτοβουλίας αλλά μόνο εάν συνδέεται με κάποια τοποθεσία. Δεύτερον, ναι, υπάρχει μια ε, διαδικασία προεπιλογής που είναι εθνική και εκεί αφήνουμε πολύ μεγάλη ελευθερία. Όμως θα υπάρξει μια ε, φόρμα, μια αίτηση η οποία θα είναι πολύ συγκεκριμένη ε, και θα δίνεται στα κράτη-μέλη. Επίσης είπαμε ότι κάθε χρονιά μπορεί να υπάρξει μία προεπιλογή το πολύ δύο ε, τοποθεσιών. Επίσης, ε, η Επιτροπή Επιλογής ε, θα αποτελείται από ανεξάρτητους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες. 12 μιλής ε, θα είναι η Επιτροπή, Τέσσερα μέλη θα έχουν οριστεί από το Κοινοβούλιο, τέσσερα από την Κομισιόν, τέσσερα από το Συμβούλιο. Τώρα, το κάθε θεσμικό όργανο έχει δικούς του κανόνες βάσει των οποίων θα επιλεγούν τα τέσσερα αυτά άτομα που θα συμμετάσχουν ε, το σημαντικό πάντως είναι ότι θα πρέπει να είναι, και αυτό είναι το πιο ουσιώδες, είναι ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης από πλευρά κρατών μελών, η πρότασή μας δεν ε, προϋποθέτει ότι θα δοθούν χρήματα ε, σε εθνικό επίπεδο. Αυτό όμως που είναι προαπαιτούμενο είναι η σωστή διαδικασία της ε, διαδικασίας προεπιλογής. Εμείς προτείνουμε η διαδικασία αυτή να είναι ε, ευέλικτη και θέλουμε πραγματικά να είναι όσο γίνεται πιο ευέλικτη και απλή η διαδικασία. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία προεπιλογής αποτελεί ένα κόστος για τα κράτη-μέλη, όντως. Αλλά αυτό είναι το μόνο κόστος στην ουσία. Um, Υπήρξε και ένα ερώτημα σχετικά με τις δεσμεύσεις των κρατών μελών. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι το πλεονέκτημα μιας εθνικής διαδικασίας προεπιλογής είναι ότι δίνουμε και ένα ρόλο στα κράτη-μέλη και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να ε, προχωρήσουν αυτή την προεπιλογή έτσι ώστε να βρουν τις ε, τοποθεσίες οι οποίες είναι πιο προσφυλείς σε αυτές. Όσον αφορά τώρα τα υλικά ε, ε, κίνητρα για τις ε, περιοχές αυτές, μετά από συζητήσεις απεφασίστη ελλείψη συνενέσεως μεταξύ των κρατών μελών, να αφήσουμε το θέμα αυτό όσο γίνεται πιο ανοιχτό και εν πάση περιπτώσει στα κράτη-μέλη. Τέλος, όσον αφορά την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, Βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι ίδιες οι τοποθεσίες μέσω προτινόμενων ε, δραστηριο... εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οπωσδήποτε θα προβάλλουν και θα, θα προωθήσουν από μόνες τους ε, τον διαπολιτισμικό διάλογο. Και επίσης σε επιχειρησιακό επίπεδο είπαμε ότι θα υπάρξει δικτύωση μεταξύ των τοποθεσιών αυτών και επομένως μπορεί να υπάρξει πρόθεση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των ιδίων των τοποθεσιών αυτών που θα έχουν το σήμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Άντσμπανς για την απάντησή σας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και την εξέταση του σημείου 5. Και βεβαίως θα επανέλθουμε στη συνεδρία των συντονιστών για να δούμε ποιος θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως. Θα έπρεπε να είχαμε παρουσίαση από τον Μιχελάνχαλ Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ, αλλά όπως σας είπα στην αρχή της συνεδρίασης, ε, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μεταξύ μας και επομένως αναβάλλεται. Επομένως νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας. Θα έχουμε συνάντηση των συντονιστών, συνεδρίαση των συντονιστών. Είχαμε πει στις 5 να γίνει συνεδρίαση των συντονιστών, αλλά δεν ξέρω. Κοιτάξτε, λέει ο Πρόεδρος, εάν δεν έχετε πρόβλημα, μπορούμε να αρχίσουμε τη συνεδρία των συντονιστών σε πέντε λεπτά. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν, πέντε λεπτό και να συνεχίσουμε αμέσως μετά με τους συντονιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνεδρίασή μας σε πέντε λεπτά συντονιστές.